και περαιτέρω εγγραφά βρίσκονται στην ειδική ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος ε, διαβίβασε τους ε, διορισμούς στην Επιτροπή Αναφορών και θα οργανωθεί μια σχετική ακρόαση των υποψηφίων. Ο συνάδελφος Βιέργια επί του κανονισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέμα κανονισμού. Συνήθως πριν ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες ακούγονται κόδωνες στο Κοινοβούλιο. Ε, πολλοί συνάδελφοι δεν ήσαν παρόντες στις ψηφοφορίες γιατί δεν ακούστηκαν τα κουδούνια στα γραφεία και στους διαδρόμους. Ε, η φήμη είναι ότι αυτό έγινε για να μην ενοχληθεί ο κύριος Γιούγκερ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε για ποιο λόγο κάποιοι συνάδελφοι ουσιαστικά εμποδίστηκαν από το να ψηφίσουν χτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριβιές. Δεν είστε ο μόνος ο οποίος αποτάνθηκε στις υπηρεσίες του σώματος σε σχέση με τον λόγο θέμα. Θα ήθελα τώρα να, σας χαιρετήσω, να χαιρετήσω στην Ολομέλεια τον κύριο Γιώργο Τσερετέλη, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής ε, Συνδιάσκεψης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να τον καλωσορίσουμε εδώ στο βήμα. Είναι μια τιμή για μας που σας καλωσορίζουμε εδώ και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ε, συζητήσεις στο Κοινοβουλίο, στο Και τώρα θα περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Ε, χρειάζεται μια απόλυτη πλειοψηφία για τις περισσότερες ψηφοφορίες. Τροπολογία Α. Α, συγγνώμη, τροπολογία Α. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται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 έχει κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την 1079. Όχι, τότε απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 1079 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 963 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Διαδικαστικό. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Thank you, Mr. President. Uh, I'd like to ask you to go slow. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μιλάτε λίγο ε, πιο αργά γιατί η διερμηνία φτάνει με λίγη καθυστέρηση και όσοι δεν κατανοούμε γερμανικά δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Όλοι λοιπόν θα επιβραδύνουμε. Λοιπόν, 964 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 902 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρινεται κατά Καταπίπτει 138-991 περ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 999 ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Κατά τα άλλα, αρκεί μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν μπορεί να γίνει εδώ εξέγερση, εάν έχετε την εντύπωση ότι έγινε κάποιο λάθος. 266 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1105 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 269 καταπίπτει. 1106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 270 καταπίπτει. Συνεπώς 1107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 993 συνεπώς καταπίπτει. Και πάμε στην 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1032 καταπίπτει, Συνεπώ, 1034 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 1033 καταπίπτει 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 1036 καταπίπτει και περνάμε στη 1113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1035 πίπτη 1264 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 999 συνεπώς πίπτη 522 υπέρ. Κατά υπέρ απορρίπτεται. 554 υπέρ. Επαλήθευση για την 522. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 554 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 434 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 435 υπέρ. Επαλήθευση για την 434. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 435 πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 436 πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα θα έρθουμε στο 1β, τροπολογία 2, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 909 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 996 καταπίπτει 262 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 263 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1201 με ονομαστική ψηφοφορία έρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι ψηφίσατε όλοι πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 989 και 280 καταπίπτουν. 559 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 912 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 1001 καταπίπτει. Συνεπώ. 1002. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται 699 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι 560 και οι 1000 συνεπώς το πρώτο τμήμα συνεπώς καταπίπτουν 2 ε, 3 ε, ηλεκτρονική ε, ονομαστική ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Πέραση ψηφοφορίας Εγκρίνεται. 1077 υπέρ κατά απορρίπτεται. 998 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1080 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1081 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 984 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1045 περ κατά αποχές απορρίπτεται 1203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 1003 καταπίπτει 1206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Υπάρχει παρανόηση για το 1206, διαφωνία όχι. 1209, 1029, ε, συγγνώμη, υπέρ. Η 1029 καταπίπτει, λέει ο πρόεδρος. 1030, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1027, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να γίνει επαλήθευση. Για τη 1027 άρχεται η ψηφοφορία. Επαλήθευση. Haben alle abgestimmt? Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Συνάδελφε Φόρμαν. Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι γελίο. Δεν μπορούμε. Είπατε πολύ γρήγορα. Οι διερμηνείς δεν προλαβαίνουν. Δεν σας προλαβαίνουν. Πρέπει να πηγαίνετε πιο αργά. Ε, μας ενδιαφέρει. Πρέπει να ψηφίσουμε σωστά τον προϋπολογισμό. Also, nochmals, meine Damen und Herren, ich werde mich... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ε, ακούστε συνάδελφε, γιατί άμα δεν με ακούσετε τότε είναι που δεν θα καταλάβετε τίποτε. Εγώ προσπαθώ, ακούω ότι σήμερα η διερμηνία στα αγγλικά είναι πιο αργή από ό,τι συνήθως. Η 1027 απορρίφθηκε, 561, ονομαστική, άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Ονομαστική ψηφοφορία η 1000 CP2. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 1050 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τίτλος 3, συνολικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Είναι ψηφοφορία 4. Πέρας. Δεκτές. Ε, 986 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 1229 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 987 πίπτη. 1047 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 308 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 141 141 πίπτη. 1226 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Καταπίπτει η 1048. 1082 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 927 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 988 καταπίπτει. 925 CP1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 1037 καταπίπτει. 1038 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12... Ε, ωραία, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 145 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 12.46 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Επαλήθευση. 12.46 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 12-22 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 149 καταπίπτει. 12-23 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 150 κατά πίπτη. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος 151. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 806 CP1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 153 καταπίπτει. 454 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 154 κατά πίπτη, 1263 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 616 καταπίπτει. Ε, συνολικά το κομμάτι ψηφοφορία 5 ψήφισαν όλοι ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. δεκτές. 5.39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.60 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 5.49 καταπίπτει. 1040 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 10.39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1041 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 1042 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 579 1043 ταυτόσημες ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία ε, ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτονται Ταυτόσημες 580-1044 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 12-15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 146 καταπίπτει. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 589 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1265 υπέρ κατά αποχές δεκτή 591 καταπίπτει 592 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται 1075 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται εψήφισαν όλοι Πέρας. Απορρίπτεται. 5-16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2-46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7-65 υπέρ. Α, έλεγχος 46 2.46. 2.46 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. 7,65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. 7,65. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. 3.28 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 403 υπέρ. Α, με συγχωρείτε. Η 403 έχει καταπέσει. Πάμε ο, συνολική ψηφοφορία, ψηφοφορία 6, ονομαστική άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτές. 595 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. 1061 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 1062 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1063 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1064 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1065 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1066 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1067 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1068 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τίτλος 5 Κοινοβούλιο, ψηφοφορία 7, συνολικά υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 6.28 υπέρ. Ορίστε συνάδελφε. Δεν είχε αρχίσει η ψηφοφορία, δεν ε, άρχισε σωστά. Συνολικά στην ψηφοφορία 7 δεν ήταν ονομαστική, δεν προβλεπόταν ε, ονομαστική, 628 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 636 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 6.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε στον τίτλο της ψηφοφορίας 8. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 5 ε, ελεγκτικό, ψηφοφορία 9, υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. 5 ε, ψηφοφορία 10 κοινωνική επιτροπή ε, υπέρ κατά αποχές δεκτές. Ε, επιτροπή των Περιφερειών, ψηφοφορία 11 συνολικά υπέρ κατά αποχές δεκτές. Ο διαμεσολαβητής, ψηφοφορία 12 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Ευρωπαϊκή Επόπτηση της Προστασίας Δεδομένων, ψηφορία 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, ε, εξωτερικής δράσης, ψηφορία 14 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Τροπολογία 204 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 678 κατά πίπτη 205 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 6,79 πίπτη. 6,80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 208 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6,81 πίπτη. 209 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6,82 καταπίπτει ε, εντάξει κύριε Φόρμαν, 221 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 683 καταπίπτει, 1250 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 684 και 250 καταπίπτουν. Μετά, μία τροπολογία ακόμα για τις δαπάνες έξω από το πολιετές, η 1046 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ε, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη 1046. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. Πάμε τώρα τα πιλωτικά προγράμματα, προπαρασκευαστικές δράσεις, ψηφοφορία 15 συνολικά. Ονομαστική, ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται. Όλες οι άλλες για τα πιλωτικά και τα προπαρασκευαστικά καταπίπτουν. Για την Προεδρία του Συμβουλίου ο κύριος Κιλικάινεν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υπέβαλε τροπολογίες στη θέση του ε, Συμβουλίου για το Δημοσιονομικό έτος 2020. Σημειώνω τις διαφορές στις θέσεις των δύο θεσμικών οργάνων σχετικά το σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 όπως το υπέβαλε η Κομισιόν. Συνεπώς, υπό την ιδιότητά μου ως Προεδρεύον του Συμβουλίου συμφωνώ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, ε, ακολουθήσει το σημείο C, παράγραφος 4 του 314 της συνθήκης για τη, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ η ψηφοφορία δεν χρειάζεται, ψηφοφορία δεν χρειάζεται εδώ και προχωρούμε. Στην έκθεση Χολμάιερ αρχίζουμε παράγραφος 1, τροπολογία 1, Χολμάιερ Ρουμπιάλ, κατά. Α, επαναλαμβάνουμε, ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 1 παρακαλώ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 2, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο καταπίπτει. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 76 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 42 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 38. Ε, Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 39. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 35. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 27 σε τρία τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το τέτοιο τμήμα καταπίπτει. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 30 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική. Ψηφίσατε όλοι. τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 59 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 62 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Πέραση ψηφοφορίας απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 θα ελέγξουμε την 63 άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 64 ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 ονομαστική, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 55 ονομαστική. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 41. Ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 37. Ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 ονομαστική. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 ονομαστική. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 15. 15 ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίες, απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 ονομαστική άρχεται ψήφισαν όλοι πέρας Απορρίπτεται 31. Ονομαστική άρχεται ψηφοφορία. 31. Ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 35 παράγραφος. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Δύο. Δεύτερο τμήμα. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης απορρίπτεται. 72 ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέραση ψηφοφορίας απορρίπτεται 19 σε τρία τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές επανάληψη ε, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Η μία πολιτική ομάδα δεν αντιδρά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας της Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Επαλήθευση για το τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Εάν 20 ε, ε, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 40 Ε, Προφορική τροπολογία. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να υποστηρίξουν την πρόταση αυτή, ανησυχούν για την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών. Το σύνολο λοιπόν της τροπολογίας λέει ότι παγώνουν όλες οι πληρωμές πιστώσεων προς την Τουρκία με εξαίρεση την βοήθεια προς την κοινωνία των πολιτών τους πρόσφυγες μέχρι το τέλος της εισβολής στην βορειοανατολική Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Να, να εξηγήσω, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, μόνο αντιρρήσεις πρέπει να εκφραστούν. Ε, ε, στέκεστε όρθια αν έχετε αντίρρηση. Πάνω από 40 συνάδελφοι δεν εγκρίνεται η προφορική. Ψηφίζομαι όπως ήταν αρχικά η 40 υπέρ. Κατά. Δεν, δεν φαίνεται το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 40 στην αρχική της μορφή. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 21 ονομαστική. Άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 16. Ονομαστική. Άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συνολικά το ψήφισμα ονομαστική άρχεται ψήφισαν όλοι Πέρασε. δεκτό προχωρούμε τώρα έκθεση Σαρβαμά Έχουμε μία ψηφοφορία για το σύνολο, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Προχωρούμε. Έκθεση Γκαρσία Μουνιός. Επίσης απαλλαγή από ε, ψήφισμα ε, υπέρ κατά αποχές δεκτό. Το ψήφισμα ε, συνολικά ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Τώρα. μια αντίρρηση, ψήφισμα για μια αντίρρηση ε, βάσει του 112 άρθρου για τις, τα φυτοφάρμακα και την επίπτωση στις μέλισσες. Ε, εδώ θα ήθελα να πω και προς τους νέους αφήστε το, την κάρτα στο μηχάνημα μέχρι να σβήσει το φως από το μηχάνημα. Μετά αν βγάλετε πιο πριν την κάρτα, χάνεται η ψήφος. Δεν ε, υπάρχει ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε ε, αποχή. Λοιπόν, ψηφίζομαι το κείμενο συνολικά. Χρειάζεται απόλυτη ε, πλειοψηφία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Ε, τιμήστε την καλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξερχόμενη της αίθουσας με το σωστό τρόπο. Ε, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, συνάδελφοι, ε, έκανα λάθος. Θέλω να δώσω στον Επίτροπο πάνω σε αυτό το θέμα το λόγο. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβουμε υπόψη μας το ψήφισμα το οποίο μόλις υιοθετήσατε. Σύμφωνα και με τη διαδικασία του κανονισμού 368 για την επιτροπολογία και σύμφωνα με τον κανονισμό 1107 Έχει υπάρξει ευνοϊκή απόφαση μέχρι τώρα για τη διαδικασία την οποία ακολουθήσουμε. Δεν θα θέλαμε να απορριφθεί μια τροπολογία η οποία προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το θέμα του κινδύνου ε, σε σοβαρό επίπεδο της, ε, μελισσο, ε, της εκτροφής μελισσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, ήταν λάθος μου λέει ο πρόεδρος προς τον Επίτροπο. Παρακαλώ, φύ, ε, εγκαταλείψτε την αίθουσα ησύχως. Όσοι δεν θέλετε να ακούσετε τις επεξηγήσεις ψήφου. Βλέπω ακόμα αρκετούς ορθίους. Θα τους αναφέρω ονομαστικά. και θα τους παρακαλέσω να ε,

Κύριε Γκάλερ. Κύριε Μακάλιστερ. Frau Kollegin Kalniete. Herr Kollege Weber. Kollegin Metzola. Herr Kollege McAllister, Herr Kollege Gahler, Herr Kollege Weber, Frau Kollegin Kalniete herr kollege danjean! so dann beginnen wir mit den stimmerklärungen. Θα ξεκινήσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου. Καταρχήν, των δύο συναδέλφων η έκθεση. Χολμάια Ρουμπιάλ, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2020, όλα τα τμήματα. Ο συνάδελφος Λούντγκρεν. Eh, Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Μόλις ψηφίσαμε για το Γενικό Προϋπολογισμό εμείς καταψηφίσαμε την πρόταση. Αυτό σημαίνει για μας ότι τεράστιες ποσότητες πιστώσεων ε, ξοδεύονται χωρίς κανένα λόγο και δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να μειωθεί ο προϋπολογισμός ενώ εσείς ζητάτε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Ε, χαμένα πάνε όλα αυτά τα λεφτά στα διάφορα θεσμικά όργανα το ελεγκτικό συνέδριο μας αποκάλυψε ότι το Συμβούλιο Υπουργών χρησιμοποίησε ένα εκατομμύριο κορώνες σουηδικές για 4.000 φιάλες καμπανίτι ίνου. Συνεπώς λοιπόν αυτά όλα πληρώνονται όπως και άλλες ε, δαπάνες με χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου και 300.000 για έπιπλα ακριβών σχεδιαστών. Frau Kollegin McGuinness, Herr Kollege Karas. So, vielen Dank, Herr Kollege Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η συνάδελφος να εξηγήσω ότι εγώ επισκέφθηκα την ε, Παλαιστίνη ο ίδιος και θα πρέπει να διαπιστώσουμε τις επιπτώσεις που έχουν οι, ε, τα κατεχόμενα στην χώρα. Ε, τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την UNRWA υπάρχει μια υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών όσον αφορά την εκτίμηση της κρίσης στην ε, Μέση Ανατολή και αυτή, ε, αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους πολίτες που, βρίσκονται, ε, που ζουν, διαβιούν στο, στην Παλαιστίνη και στη Γάζα. Ε, επίσης, ήρθα σε επαφή με τις οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα έχουν επαφέ με την UNRWA. Ε, σε σχέση με τα προγράμματα προσφύγων, με τα παιδιά κλπ. υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα και εμείς δεν θα έπρεπε να αυξήσουμε τον ε, προϋπολογισμό γιατί με τον τρόπο αυτό υπονομεύουμε την ε, κατάσταση ε, των, ανθρώπων στην Παλαιστίνη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον συνάδελφο κύριο Σιόλος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλερ. Ο κύριος Βάιμερς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι κατά αυτού του προϋπολογισμού γιατί πραγματικά βρήθη από σπατάλες τα βασικά, το βασικό, τα βασικά, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα. Ο λόγος για τον οποίο μιλώ στα γερμανικά είναι ότι θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία προκειμένου να πω στον κύριο Μάνφρετ Βέμπερ, τον πρόεδρο της ΕΛΚ, ε, να του πω το εξή ερώτημα. Ασφαλώς κύριε Βέμπερ, εσείς ως συντηρητικός θέλετε να διατηρήσετε τη φορολόγηση σε ένα λογικό επίπεδο. Αλλά τότε γιατί κάνετε αυτό το δώρο του εισιτηρίου το, στο Interrail γιατί εδώ αποτυγχάνει τόσο το μοντέλο του σοσιαλισμού οι φορολογούμενοι στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αποφεληθούν εάν βρίσκατε εσείς μια πανάκια έναντι αυτού του τύπου εφαρμογής του σοσιαλισμού. Ο κύριος ε, Πόσπιστήλ. Ευχαριστώ. Εγώ ψήφισα το σχέδιο προϋπολογισμού γιατί έχει πολλά θετικά. Το σημαντικό είναι η Frontex για μας. Περισσότερα κονδύλια για τη Frontex και για το Erasmus επίσης, που είναι σημαντικότατο πρόγραμμα που στηρίζει την κινητικότητα των νέων και την εκπαίδευση που είναι έμεσος τρόπος καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Και αυτό που είναι θετικό είναι ότι το 1 πέμπτο του προϋπολογισμού ε, αφιερώνεται σε περιβαλλοντικά προγράμματα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εδώ συζητούμε αν ε, παλεύει για την, ενάντια στην κλιματική αλλαγή η Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός αποδεικνύει πως ναι, ε, παίρνουμε μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής. Στηρίζω τον προϋπολογισμό λοιπόν και πιστεύω ότι στο τέλος οι συζητήσεις θα οδηγήσουν στην έγκριση του από τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κάρθη. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την συγκεκριμένη έκθεση, διότι αυτά είναι στρατιωτικά θέματα και η χώρα μου, η Ιρλανδία, είναι μια θα έλεγα δέσμευτη ε, και ουδέτερη σε τέτοιου είδους θέματα και γι' αυτό δεν θέλω να πιέζεται η χώρα μου προς ε, μια δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού. Ευχαριστώ συνάδελφε Κάρθη, συνάδελφος Χιόιτροβα. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι, αγαπητοί πολίτες που παρευρίσκεστε. Εγώ στήριξα το σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 γιατί περιλαμβάνει σημαντικότατες λύσεις, λύσεις που στηρίζουμε. Το πρόγραμμα Εράσμους για την εκπαίδευση των νέων και την κινητικότητα των νέων αυτό το χρειαζόμαστε. Τα τελευταία έξι χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε ε, και δημιούργησε 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάρη στον προϋπολογισμό για ανεργούς νέους. Κάποιες ε, προτάσεις ε, δικές μας δυστυχώς απερίφθησαν ε, για παράδειγμα που αφορούσαν την κοινή αγροτική πολιτική που κάποιοι ήθελαν να σταματήσουν. Αυτό απερίφθη. Ευτυχώς απερίφθη γιατί χρειαζόμαστε αυτή την πολιτική. Και εμείς σταματήσαμε ε, να χρηματοδοτούμε και να προωθούμε τις προενταξιακές ε, πραγματεύσεις με την Τουρκία. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατία στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σιόιντροβα. Δεν ήθιστε να έχουμε εκφράσεις επί, επικο, δοκιμασίας ή αποδοκιμασίας. Όπω και οι συνάδελφοι του Εθνικού Συναγερμού καταψήφισαν την τροπολογία 37 τη έκθεσης Χολμάγερ που κατέθεσαν οι ομάδες της Άκρα Αριστεράς ε, γιατί ζητούν την κατάργηση τη κοινή αγροτική πολιτική. Μπορεί να ασκήσει κανεί ε, κριτική στην ΚΑΠ και μπορεί να την αντικαταστήσει κάποτε με ένα άλλο σύστημα όπου το κάθε κράτο θα είναι υπεύθυνο για τη δική του γεωργία. Προ στιγμή όμω η κοινή αγροτική πολιτική υπάρχει και στηρίζεται πολιτικά. Το μόνο που μπορούμε βαχυπρόθεσμα να κάνουμε είναι να την συντηρήσουμε εποφελούμενοι από την εξελίξη διαπραγμάτευση για να την βελτιώσουμε και θα πρέπει επίσης να βάλουμε ένα ανώτατο όριο στα χρήματα που δίδονται στις μεγάλες καλλιέργειες έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες γεωργικές επιχειρήσεις σε ανθρώπινο μέγεθος που είναι χαρακτηριστικό άλλωστε και της γαλλικής κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λεμπρετόν. Ακολουθεί συνάδελφος κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι υπερψήφισα τον προπολογισμό του προσεχούς έτους για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι αρκετά φιλόδοξος σε σχέση με συγκεκριμένα προγράμματα ε, όπως είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Βεβαίω εδώ χρειάζονται ε, περισσότερα κονδύλια προκειμένου να αποφεληθούν ε, και οι πολίτες στην, στην περιφέρεια της Υπέθρου. Η τροπολογία υπαριθμών 20, την οποία